Σε ό,τι αφορά τώρα τις ασυλίες, η κυρία Χαουτάλα διορίζεται εισηγήτρια για την άρση ασυλίας ε, του Μπελακόβατ. Σε ό,τι αφορά τώρα τις κατοξιδότητες πράξεις και τις ε, εκτελεστικές πράξεις, Λουκμάστρουμ ε, ορίζεται εισηγητής για τον εφαρμοστικό κανονισμό της Κομισιόν που θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες για να εφαρμοστούν ορισμένες διατάξεις του κανονισμού του Συμβουλίου 2007 κάθετος 2009 για το ε, σήμα, το εμπορικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνήσαμε να ζητήσουμε αξιολόγηση του κόστου της μη Ευρώπης από τη γνώμα ΔΕΛΤΑ EPRS σε σχέση με την ε, έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας για τους κανόνες αστικού δικαίου για τη ρομποτική. Και τέλος συμφωνήθηκε να ζητήσουμε μελέτη αντικτύπου για την πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου για μια ανεκτή αποτελεσματική ευρωπαϊκή διοίκηση. Αυτά ως προς τις ανακοινώσει και μπορούμε να συνεχίσουμε τώρα με το σημείο 9, η παρουσίαση της ε, μελέτης του Τμήματος Πολιτικής ε, ΓΑΜΑ για τα ατυχήματα, τα διασυνοριακά ατυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τον πιθανό αντίκτυπο των αυτοκινήτων χωρίς ε, οδηγό. Η παρουσίαση θα γίνει από τον κύριο Τόμας Κάντνερ, Γκρατσιάνο, από το Πανεπιστήμιο της Γενέβης. Σας καλωσορίζω και θέλω να σας δώσω το λόγο. Thank you very much. I was... Ευχαριστώ πολύ μου είπαν ότι μπορώ να καθίσω και όρθιος. Τα αυτόνομα συστήματα οδήγησης για τα αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό εξέλιξη. Στο μέλλον αυτά τα συστήματα μπορούν να γίνουν ε, ε τόσο εκτεταμένα που ε, τελικά να μην χρειάζεται καν οι άνθρωποι να οδηγούν. Εάν αυτά τα αυτόνομα συστήματα αποτύχουν, ενδέχεται να υπάρξουν ατυχήματα. Εάν ένα ατύχημα συμβεί στο εξωτερικό, ε, ή τα οχήματα είναι ταξινομημένα ε, στο εξωτερικό ή τα άτομα αυτά διαμένουν στο εξωτερικό, τότε πρέπει να δούμε ε, σε ποιο δικαστήριο θα πρέπει να προσφύγει κανείς και ποιο δίκαιο ισχύει για να καθορίσουμε την αστική ευθύνη του οδηγού, του κατόχου, του κατασκευαστή ε, του αυτοκινήτου ή του κατασκευαστή της ελαττωματικής νέας τεχνολογίας. Σήμερα εξετάζουμε κατά πόσο οι κανόνες ε, του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που διέπουν και καθορίζουν μάλλον την διεθνή δικαιοδοσία και το εφαρμοστέο δίκαιο καλύπτουν επακριβώς ε, διασεμεριακά ατυχήματα τα οποία προκαλούνται από ελαττωματικές νέες τεχνολογίες ή εναλλακτικά κατά πόσο θα πρέπει να τροποποιηθούν και να προσαρμοστούν. Το θέμα αυτό μπορεί να φανεί καλύτερα αξιοποιώντα ένα παράδειγμα με βάση το νομολογία των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων. Μία οικογένεια που, για παράδειγμα, ζει στη Γαλλία, ε, παραθερίζει σε μια άλλη ε, χώρα, για παράδειγμα στην Ισπανία. Οδηγούν δύο ε, οχήματα, το ένα πίσω από το άλλο, σε έναν ισπανικό αυτοκινητόδρομο. Ο γιος που οδηγεί το μπροστινό όχημα ε, πλησιάζει σε μία αριστερή στροφή. Προκειμένου να ε, προσπεράσει ένα φορτηγό, πηγαίνει στην αριστερή λωρίδα και ξαφνικά ε, παρατηρεί ένα ΣΕΑΤ Κόρδοπα το οποίο έχει μείνει ακινητοποιημένο στην αριστερή λωρίδα μετά από ένα τύχημα. Ο νεαρός λοιπόν πατάει φρένο και έτσι αποφεύγει την σύγκρουση με το ισπανικό όχημα. Ωστόσο ο πατέρας του δεν καταφέρει να σταματήσει εγκαίρως και έχουμε σύγκρουση των δύο οχημάτων της οικογένειας. Ο γιος ε, τραυματίζεται σοβαρά και χάνει την ικανότητα εργασίας για την υπόλοιπη ζωή του. Και τα δύο οχήματα και αυτό που οδηγεί ο πατέρα και αυτό που οδηγεί ο γιο είναι ταξινομημένα και ε, ασφαλισμένα στη Γαλλία. Το ΣΕΑΤ, το οποίο δεν ε, έχει συμμετάσχει στη σύγκρουση, ε, είναι ταξινομημένο στην Ισπανία. Α υποθέσουμε τώρα ότι η σύγκρουση αυτή προκλήθηκε είτε επειδή ο πατέρα αμελώ καθυστέρησε να φρενάρει ή επειδή υπήρχε ε, στο όχημα του πατέρα μια ε, συσκευή αυτόνομης οδήγησης που ήταν αλλατοματική. Ο γιος ε, αξιώνει αποζημίωση για σωματική βλάβη και ε, απώλεια εισοδήματος από τον, την ασφαλιστική εταιρεία του πατέρα, το οποίο συμβαίνει συχνά. Ε, βάσει του κανονισμού Βρυξέλλες 1 που ισχύει σε 27 κράτη-μέλη, ε, ο ενάγων έχει τη δυνατότητα να, ε, να προσφύγει ε, στο κράτος μέλος όπου δράζεται ο ασφαλιστής, για παράδειγμα στη Γαλλία, ή εκεί που έγινε το ατύχημα, στο δικό μας παράδειγμα Ισπανία, ή στα δικαστήρια του κράτους όπου διαμένει μόνιμα το θύμα. Στο δικό μας παράδειγμα, Γαλλία. Οι κανόνες δικαιοδοσίας ε, που ε, αναφέρονται στον κανονισμό Βρυξέλλες 1 ισχύουν ανεξάρτητα από την αιτία του ατυχήματος. είτε πρόκειται για ανθρώπινο σφάλμα ή τεχνολογικό ελάττωμα. Επομένως, τέτοιοι κανόνες μπορούν να ισχύσουν και για ατυχήματα που προκαλούνται από ελαττωματικές νέες τεχνολογίες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το δίκαιο που εφαρμόζεται για τα τροχαία ατυχήματα καθονίζεται από ένα από τα δύο συστήματα διεθνούς ιδιωτικού δικαίου που υπάρχουν, ανάλογα με τη χώρα στην οποία ε, γίνεται η προσφυγή. Είτε βάσει του κανονισμού Ρώμη 2, είτε με βάση τη σύμβαση της Χάγης 1981 για το εφαρμοστέο δίκαιο σε ό,τι αφορά τα τροχαία ατυχήματα. Η σύμβαση του 1971 της Χάγης ε, κυριαρχεί επί του κανονισμού Ρώμη 2 για ε, υποθέσεις ε, ενώπιον δικαστηρίου σε κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι συμβαλόμενο μέρος στη Σύμβαση της Χάγης. Από τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 13, σχεδόν τα μισά δηλαδή, είναι συμβαλόμενα μέρη της Σύμβασης της Χάγης, συμπεριλαμβανομένης και της Γαλλίας και Ισπανίας. Τα δικαστήρια για των δύο αυτών χωρών, επομένω, θα ε, καθορίσουν το εφαρμοστέο δίκαιο βάσει των κανόνων τη Σύμβαση τη Χάγη. Σύμφωνα με τη συμφωνία τη Σύμβαση της Χάγης, η αστική ευθύνη κατόπιν τροχαίου ατυχήματο ε, διέπεται κατά βάση από το δίκαιο της χώρας στο οποίο, ε, στην οποία λαμβάνει η χώρα το ατύχημα. Στο δικό μας παράδειγμα, ισπανικό δίκαιο. Ωστόσο, όταν έχουμε πολλαπλά οχήματα, που εμπλέκονται στο ατύχημα, ε, τότε ισχύει ε, το δίκαιο του κράτους ταξινόμησης, εάν όλα τα οχήματα έχουν ταξινομηθεί στο ίδιο κράτος. Επομένω, αυτή η εξαίρεση εξαρτάται από το πού έχουν ταξινομηθεί τα οχήματα που εμπλέκονται στο ατύχημα. Ακόμα και αν το άτομο που είχε υποστεί τη σωματική βλάβη και ε, το άτομο που υποτίθεται ότι είναι υπεύθυνο έχουν την έδρα τους στο ίδιο κράτος. Για παράδειγμα, πατέρας και γιος και οι δύο στη Γαλλία. Στο δικό μας σενάριο, βάσει τη Σύμβαση της Χάκη, το εφαρμοστό δίκαιο εξαρτάται από το κατά πόσο τα οχήματα που συμμετέχουν και εμπλέκονται στο ατύχημα είναι όλα ταξινομημένα στο ίδιο κράτος μέλος. Τα οχήματα του πατέρα και του γιου έχουν ταξινομηθεί στη Γαλλία, ενώ το ΣΕΑΤ έχει ταξινομηθεί στην Ισπανία. Σύμφωνα με την ομολογία των 100 μελών ε, των συμβαλωμένων μερών της Σύμβασης της Χάγης, εάν ένα άλλο όχημα, όπως το ΣΕΑΤ στη δική μας περίπτωση, ενδέχεται να ήταν η αιτία του ατυχήματος, τότε θεωρείται ότι εμπλέκεται στο ατύχημα. Ως εκ τούτου, στο, στη δική μας περίπτωση δεν έχουν ταξινομηθεί όλα τα οχήματα στο ίδιο κράτος, επομένως εφαρμόζεται το ισπανικό δίκαιο, καθότι ήταν ο τόπος ε, που έλαβε χώρα το ατύχημα. Σε ό,τι αφορά το δικό μας ζήτημα, λοιπόν, θεωρούμε ότι οι συνδετικοί παράγοντες που χρησιμοποιούνται στην σύμβαση της Χάγης για να καθορίσουμε το εφαρμοστό δίκαιο, δηλαδή τόπος του ατυχήματος ή χώρα ταξινόμησης των οχημάτων, δεν εξαρτώνται από την αιτία του ατυχήματος. Οι κανόνες που θεσπίζονται από τη Σύμβαση της Χάκης μπορούν λοιπόν να εφαρμοστούν και σε περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων που προκαλούνται από λατωματικές νέες τεχνολογίες. Αυτά είναι τα καλά νέα για σήμερα. Τώρα τα άσχημα νέα. Στο παράδειγμά μας είναι ότι ε, οι νόμοι αστικής ευθύνης, ουσιαστικής ε, ε, διαφέρουν από το, σημαντικά μάλιστα από τη μία χώρα στην άλλη. Ενώ στο γαλλικό δίκαιο, όπου και οι δύο εδρεύουν, στη δική μας περίπτωση, ισχύει η αρχή της πλήρους αποζημίωσης. Από την άλλη όμως, το ισπανικό δίκαιο προβλέπει αποζημίωση ε, που έχει συγκεκριμένα όρια, τα λεγόμενα μπαρέμους. Και μάλιστα σε ό,τι αφορά την απώλεια εισοδήματο, αυτή η αποζημίωση είναι πολύ χαμηλότερη ε, σε σχέση με την ζημία που όντω υπέστη ο νεαρό στην περίπτωσή μα. Εφόσον και τα δύο μέρη ε, της υπόθεσης εδρεύουν στην Γαλλία, και ότι η παρουσία του στην Ισπανία ήταν πολύ σύντομη, το αποτέλεσμα μπορεί να θεωρηθεί άδικο για το δίκαιο και απροσδόκητος, ε, απροσδόκητο λαχείο, αν θέλετε, για την ασφαλιστική ε, του πατέρα. Αυτή είναι μία από τις αρκετές σημαντικές διαφορές μεταξύ των ε, νόμων που ισχύουν σε επιμέρους κρατών μελών σε επιμέρου Στη δική μα περίπτωση, το εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ισπανικό, ανεξάρτητα από το κατά πόσο ε, προσέφυγε ο ε, ενάγων σε γαλλικό-ισπανικό δικαστήριο, γιατί και οι δύο εφαρμόζουν τη Σύμβαση τη Χάγη. Όμω, πώ θα ήταν τα πράγματα εάν η οικογένεια αυτή ε, διέμενε μόνιμα στη Γερμανία αντί για τη Γαλλία. Η Γερμανία είναι ένα από τα 15 κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν είναι συμβαλόμενο μέρο στη Σύμβαση τη Χάγη. Ενώπιον των Γερμανικών Δικαστηρίων, το εφαρμοστείο δίκαιο έτσι καθορίζεται από τον κανονισμό Ρώμη 2. Με βάση τον κανονισμό ΡΟΜΗ 2, η αστική ευθύνη κατόπιν τροχαίου ατυχήματο επίση ε, καταρχήν διέπεται από το δίκαιο τη χώρα ε, στην οποία έλαβε χώρα το ατύχημα. Όμω, εάν το δικαίωμα που θεωρείται, το, το άτομο που θεωρείται υπεύθυνο και το άτομο που υπέστη την ε, ζημία και οι δύο διέμεναν μόνιμα στην ίδια χώρα της, κατά τη στιγμή της, του ατυχήματο, τότε ο, ο κανονισμό ΡΟΜΗ 2 ισχύει για την εφαρμογή του δικαίου της ε, χώρας αυτής αντί για το δίκαιο της χώρας ε, στην οποία έλαβε χώρα το ατύχημα. Γιατί και τα δύο μέρη πρέπει να υποστούν τις συνέπειε του ατυχήματος στην ίδια χώρα και υπάρχει πολύ στενότερος δεσμός με αυτή τη χώρα παρά με τη χώρα του ατυχήματος όπου τα μέρη, οι διάδικοι ε, πέρασαν μόνο ένα μικρό χρονικό διάστημα. Επομένως, στη δική μας περίπτωση Εάν ε, τα, πατέρας και γιος διέμεναν μόνιμα στη Γερμανία, τότε τα γερμανικά δικαιώματα θα εφαρμόσουν το γερμανικό και όχι το ισπανικό δίκαιο και ο γιος θα λάβει πλήρη αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη, ε, συμπεριλαμβανομένης και πλήρους αποζημίωσης για την ε, διαβίου απώλεια εισοδήματος. Και πάλι εδώ οι συνδετικοί παράγοντες ε, που αξιοποιούνται από τον κανονισμό Ρώμη 2, δηλαδή το, ο τόπο ατυχήματο η ε, συνήθις, ο συνήθι τόπο κατοικία στην ίδια χώρα, δεν εξαρτώνται από την αιτία του ατυχήματο και έτσι επίσης μπορούν να εφαρμοστούν σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το ατύχημα ε, προκλήθηκε από νέε τεχνολογίε. Ωστόσο, Από τα προηγούμενα σενάρια προέκυψε ότι οι συνδετικοί παράγοντες στον Ρώμη 2 είναι πιο σύγχρονοι και πιο κατάλληλοι ε, για τα δύο μέρη σε ένα ατύχημα και πιο συγκεκριμένα για το θύμα από ότι οι κανόνες ε, της σύμβασης της Χάγης. Μία πρώτη επίπτωση, ένα πρώτο συμπέρασμα είναι ότι η σύνδεση μεταξύ της σύμβασης της Χάγης του 71 και του κανονισμού Ρωμιδίου θα πρέπει να τύχει επαναδιαπραγμάτευσης και επαναπροσδιορισμού. Το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού Ρώμη 2 θα μπορούσε, για παράδειγμα, να επεκταθεί για να καλύψει όλες τις περιπτώσεις στις οποίες και ο ενάγων και ο εναγόμενος εδρεύουν σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα βρείτε και μια πιο συγκεκριμένη πρόταση για μια τέτοια τροποποίηση στη σελίδα 28 της μελέτης μας. Εάν ένα σενάριο, σαν αυτό στη δική μας περίπτωση, έχει ε, προκληθεί από ελαττωματική τεχνολογία, το θύμα, στη δική μας περίπτωση ο νεαρός, μπορεί επίσης να ε, καταθέσει αγωγή κατά του κατασκευαστή του ελαττωματικού οχήματος που προκάλεσε το ατύχημα ευθύνη που συνδέεται με τα προϊόντα λοιπόν ε, θα λάβει κατά πιθανότητα μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτό το τομέα. Ας πούμε ότι το όχημα που οδηγούσε ο πατέρας ε, με την ελαττωματική τεχνολογία είχε κατασκευαστεί στη Σουηδία. Με βάση τον κανονισμό, με ε, Βρυξέλλες 1, το άτομο που υπέστη τη ζημία έχει το δικαίωμα να καταφύγει στα, δικαιώματα, στα δικαστήρια του κράτους μέλους ε, της Σουηδίας, όπου εδρεύει ο κατασκευαστής, ή στα δικαστήρια του τόπου που έλαβε χώρα το ατύχημα, σε αυτή την περίπτωση Ισπανία. Από την άλλη μεριά, τα δικαστήρια του κράτους όπου εδρεύει το θύμα, εδώ Γαλλία, έχουν δικαιοδοσία μόνο για την αγωγή κατά του κατασκευαστή του οχήματος υπό τον Βρυξέλλες 1, εάν ο κατασκευαστής του οχήματος είχε ε, αποκτήσει ασφάλεια αστικής ευθύνης που καλύπτει ε, και τρίτους και επιτρέπεται και ε, απευθείας αγωγή κατά του κατασκευαστή. Στην πράξη βλέπουμε ότι τα θύματα τροχαίων εποφελούνται σε μεγάλο βαθμό της δυνατότητας άμεσης αγωγής κατά του ασφαλιστή του αναγόμενου και συνήθως προτιμούν να προσφέρουν στα δικαστήρια της χώρας τους. Αυτό επιβεβαιώνεται από πάρα πολλές υποθέσεις. Δεύτερη συνέπεια της ε, μελέτης μας είναι ότι θα πρέπει να εισαγάγουμε, για παράδειγμα, ε, σε συγκεκριμένες οδηγίες ασφάλισης ε, κινητήρων, ε, μία ε, υποχρέωση για τους ε, κατασκευαστές αυτοκινήτων να αποκτούν τέτοια σύμβαση που να καλύπτει και αστική ευθύνη για τα θύματα τροχιών ατυχημάτων και μια δυνατότητα άμεσης αγωγής κατά του ασφαλιστή του κατασκευαστή. Εάν εισαχθούν και, τα δύο, και οι δύο αυτές διατάξεις, τότε τα άρθρα 13.2 και 11.1β του κανονισμού Βρυξέλλες 1 θα ισχύσουν και το θύμα μπορεί να ε, ε, καταθέσει αγωγή κατά του ασφαλιστή του κατασκευαστή στα δικαστήρια της χώρας του στην οποία διαμένει. Στο δικό μας παράδειγμα, ο νερός θα μπορούσε να αξιώσει αποζημίωση ε, από τον κατασκευαστή του οχήματος του πατέρα του ενώπιον των γαλλικών δικαστηρίων στην χώρα διαμονής του. Οι κανόνε αστική ευθύνη των κρατών μελών διαφέρουν σημαντικά λοιπόν, όχι μόνο σε ό,τι αφορά του ε, τους όρους της αστικής ευθύνη, τον κύκλο των ατόμων που επωφελούνται από την αυστηρή αστική ευθύνη και τα ποσά που επιδικάζονται, αλλά και σε ό,τι αφορά τον χρονικό περιορισμό που ισχύει ε, για αξιώσεις εξωσωματικής αστικής ευθύνης. Έτσι, συχνά, μία τέτοια αγωγή ε, παραγράφεται υπό το εφαρμοστέο ε, ξενοδίκαιο, ενώ υπό το δίκαιο της χώρας την οποία διαμένει το θύμα θα μπορούσε ακόμα να κατατεθεί η αγωγή. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, έχουμε μόνο ένα χρόνο ε, χρονικό περιθώριο και είναι μάλιστα από τα πιο ε, σύντομα, ενώ στη Γαλλία είναι από τα πιο μακροχρόνια. Αυτό μπορεί να εκπλήξει τα, τα θύματα τέτοιων τροχιών ατυχημάτων που κινδυνεύουν να χάσουν τη δυνατότητα να καταθέσουν αγωγή υπό το ξένο δίκαιο που ε, εφαρμόζει συγκεκριμένο χρονικό περιορισμό. Αυτό θα μπορούσε να επιληθεί είτε με την επέκταση του χρονικού περιθεωρίου ε, σε επίπεδο ουσιαστικού δικαίου, το οποίο μπορεί να είναι δύσκολο όντως ε, να συμφωνηθεί στην Ευρώπη, ή κάτι το οποίο θα ήταν πιο εύκολο να υλοποιηθεί, με το να ε, εισαγάγουμε έναν αθρεστικό συνδετικό μηχανισμό σε επίπεδο διεθνούς ιδιωτικού δικαίου, με βάση το οποίο ε, μια τέτοια αγωγή παραγράφεται μόνο εάν έχει εκπνεύσει προθεσμία και υπό το δίκαιο που ε, εφαρμόζεται για την αξίωση αστικής ευθύνης και υπό το δίκαιο του κράτους ε, στο οποίο εδρεύει το θύμα, υπό τον κανονισμό Ρώμη Και θα βρείτε ακριβή πρότασή μας στην σελίδα 51 και 57 της μελέτης. Κλείνοντας, Υπάρχουν τέσσερις πιθανές ενέργειες που προτείνουμε για να βελτιώσουμε την θέση των θυμάτων των διασυνοριακών τροχιών ατυχημάτων. Πρώτον, καλύτερο συντονισμό του κανονισμού ΡΟΜΗ 2 και τη σύμβαση της Χάγης του 71 για τα τροχιά ατυχήματα. Βλέπε πρόταση για τροποποίηση του κανονισμού ΡΟΜΙ 2 στη σελίδα 28 της μελέτης. Δεύτερον, να εισαγάγουμε σε επίπεδο ουσιαστικού δικαίου υποχρέωση για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων να ε, κατέχουν ασφάλιση αστικής ευθύνης που να καλύπτει και τα θύματα τροχιών ατυχημάτων μαζί, και αυτή είναι η τρίτη πρόταση, με άμεση ε, αγωγή για τα θύματα τροχιών ατυχημάτων κατά του ασφαλιστή του κατασκευαστή. Εάν συμβεί αυτό σε επίπεδο διεθνούς ιδιωτικού δικαίου, το θύμα αυτομάτως επωφελείται ε, ε, της δυνατότητας ε, να προσφύγει σε δικαστήριο της χώρας του υπό τον κανονισμό Βρυξέλλες 1. Και δεν χρειάζεται να τροποποιηθεί αυτός ο κανονισμό. Και τέταρτη πρόταση, να εισαγάγουμε έναν ε, αθρηστικό συνδετικό μηχανισμό στον κανονισμό Ρώμη 2, με βάση τον οποίο μία ε, τέτοια ε, περίπτωση παραγράφεται μόνο εάν έχει εκνεύσει η προθεσμία και υπό το δίκαιο που εφαρμόζει την αξίωση και υπό το δίκαιο του κράτους στο οποίο εδρεύει το θύμα. Έτσι έχουμε δύο τροποποιήσεις στον ε, κανονισμό ρομι 2 και δύο τροποποιήσεις ε, στην οδηγία περί κινητήρων. Ευχαριστώ. Thank you as well, Professor, for your Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας και για τις συγκεκριμένες ε, προτάσεις που κάνατε. Ε, και τα να δω αν υπάρχουν ερωτήσεις ή παρεμβάσεις από τα μέλη. Αλλά δεν βλέπω να υπάρχουν. Αυτό σημαίνει ότι πραγματικά ήταν, κάλυψε όλο το θέμα η παρουσίασή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ σήμερα. Ε, σίγουρα θα επανέλθουμε στα θέματα αυτά μελλοντικά. Ιδιαίτερα την πρόεδρος κυρία Ντελβό η οποία προείσατε της ομάδας εργασίας για τη ρομποτική. Α, η κυρία Ντελβό θέλει να σχολιάσει. Α, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ συγκεκριμένη η παρουσίασή σας και άρα πολύ χρήσιμη για τους προβληματισμούς μας. Ε, σήμερα το πρωί είχα την ευκαιρία να κοιτάξω το γραπτό σας κείμενο. Και το ερώτημά μου είχε, ήταν, αφορούσε το θέμα της ε, ευθύνης, γιατί δεν αναφερθήκατε σε αυτό. Ε, όλες οι χώρες έχουν ένα τέτοιο μοντέλο περιφέρειας. Uh, Στη μελέτη, η, μελέτη επικεντρώνεται στο αστικό δίκαιο, άρα βασίζουμε σε κάποιες παραδοχές. Και η δική μου παραδοχή ήταν ότι θα πρέπει να είναι αυτονόητο ότι χρειαζόμαστε ένα σύστημα αυστηρή ευθύνη σε όλες τις ε, χώρες ε, μέλη για τα αυτοκινητιστικά ατυχήματα. Ε, και υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις στο αστικό δίκαιο, το Ιρλανδικό δίκαιο και το Βελγικό δίκαιο, το οποίο όμως τροποποιήθηκε. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι χρειαζόμαστε στο επίπεδο του ουσιαστικού δικαίου ένα, αυστηρό, ένα σύστημα αυστηρής ευθύνης για ζημίες που προκαλούνται από δικά ατυχήματα. Αυτό είναι φτανότητα στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην, στην ε, Ελβετία και σε πολλές άλλες χώρες. Το πρόβλημα είναι όμως ότι σε ορισμένες χώρες ο κύκλος των ανθρώπων που επωφελούνται από αυτή την ευθύνη ποικίλει. Σε ορισμένες χώρες οποιοδήποτε θύμα μπορεί να επωφεληθεί, ε, σε άλλοι επιβάτες των οχημάτων δεν μπορούν να επωφεληθούν, πρέπει να αποδείξουν την αμέλεια και σε ορισμένα συστήματα οι επιβάτες στα οχήματα το οποίο προκάλεσε το ατύχημα δεν μπορούν να αποφεληθούν από αυτή την ε, ευθύνη, την ευθύνη. Ε, άρα λοιπόν η επέκταση αυτής της έννοιας strict ε, liability για να προστατευτούν όλα τα θύματα των ε, ατυχημάτων αυτοκινηστικών είναι μια λύση για το μέλλον. Σε ορισμένε χώρες η strict liability αφορά πεζούς ή και θα έπρεπε βεβαίως να επεκταθεί σε επιβάτες των οχημάτων. Ωραία λοιπόν, υποθέτω ότι ένα τέτοιο ε, σύστημα θα ήταν ε, χρήσιμο. Στην Αγγλία και στην Ιρλανδία έχουμε άλλο σύστημα και βλέπουμε στην Ιρλανδία ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου ο δικαστής πραγματικά παλεύει να εντοπίσει σφάλματα του οδηγού προκειμένου να προστατευτούν τα θύματα αλλά αυτό καμιά φορά είναι πολύ δύσκολο. Άρα λοιπόν η έννοια αυτή, ε, strict liability, αυστηρή ευθύνη, θα έπρεπε ε, να ε, διατυπωθεί με ακρίβεια. για ένα θύμα το να αποδείξει τι ακριβώς προκάλεσε το ατύχημα είναι σχεδόν αδύνατο. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει εισαχθεί η νέα αυτή τεχνολογία, είναι αυτονόητο ότι χρειαζόμαστε αντικειμενική ευθύνη, αντικειμενική ευθύνη των κατασκευαστών και θα έπρεπε να επεκταθεί σε όλους. Σε πολλές χώρες αυτή η έννοια της αντικειμενικής ευθύνης θα άλλαζε τα πράγματα και θα ε, κάλυπτε πολλά ελλείμματα. Εάν μπορώ να προσθέσω κάτι που αφορά τις ε, περιόδους περιορισμών στην Ευρωπαϊκή συγγνώμη, ε, για οδικά ατυχήματα. Εάν έχουμε την πεποίθηση ότι η ευθύνη θα είναι, η έννοια της αντικειμενικής ευθύνης θα είναι πιο σημαντική, θα είναι σημαντικό να αστιαστούμε όχι μόνο στα οδικά ατυχήματα, ε, το κλασικό σύστημα αποζημιώσεων για τα δικά ατυχήματα, αλλά επίση να εξασφαλίσουμε ότι νέε περίοδοι παραγραφής ε, θεσπίζονται ε, εν σχέση με την πλατύτερη έννοια της ευθύνης, όπου εφαρμόζονται οι κανόνες για τα δικά ατυχήματα. Γιατί εδώ εφαρμόζονται κάποιοι, κάποιες ευρύτερες ε, διάρκειες ε, παραγραφής. Και για να προσθέσω μια τελευταία φράση. Εάν ε, προσεγγίσουμε το θέμα στο επίπεδο του Διεθνούς Ιδιωτικού Δικαίου και πούμε ότι η ανέργεια παραγράφεται μόνο εφόσον είναι, μπορεί να παραγραφεί σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και το δίκαιο στην χώρα παραμονής του θύματος ε, όπως για παράδειγμα στην Ελβετία όπου είναι ένα χρόνο, όπως και στην Ισπανία, είναι μικρό δηλαδή το διάστημα αυτά. Άρα λοιπόν το θύμα από μια άλλη χώρα και στην Τσεχία είναι πολύ σύντομο. Ε, δεν θα ε, ευνηδιαζόταν από μια τόσο σύντομη διάρκεια αλλά όταν ε, η παραγραφή στην άλλη χώρα είναι 4 ή 5 χρόνια, ε, ε, υπάρχει εδώ μια μεγάλη απόκληση. Αυτή τη στιγμή διασχίζει κανείς τα σύνορα, νομολογία είναι πολύ δύσκολο να ερμηνευθεί και αυτές ε, οι μικρές ε, περίοδο, περίοδοι παραγραφής δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε διασυνοριακές περιπτώσεις. Κάναμε μελέτες και είδαμε ε, την ομολογία την οποία αναλύσαμε και αναρωθήκαμε γιατί οι περιπτώσεις προσέφηκαν στο δικαστήριο και είδαμε ότι 25-33% των περιπτώσεων ο λόγος ήταν ότι υπό αλλοδαπό εφαρμοστέο δίκαιο η, η πράξη είχε παραγραφεί ενώ στις χώρες των θυμάτων ε, δεν ίσχυε η παραγραφή και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό έβριμα. Well, ε, Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε λοιπόν το ζήτημα αυτό. Σας ευχαριστούμε κύριε καθηγητά που ήσασταν εδώ και μας παρουσιάσατε τις γνώσεις σας. Θα συνεχίσουμε. Θα έπρεπε να συνεχίσουμε με το σημείο 11. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Ντυρά, που είναι εισηγητής, δεν είναι εδώ. Θα έρθει αργότερα. Επομένως, πάμε στο σημείο 12. Έχουμε την ε, μελέτη των εκφραστικών ε, μέτρων και την εξοδότηση πράξεων. Σίλια Βίξτρομ είναι η συγγήτρια. Όχι ότι θα ήταν εδώ. Όμως, να σας ανακοινώσω ότι οι συντονιστές έχουν διορίσει την κυρία Βίξτρομ ως εισηγήτρια καθώς ήταν η εισηγήτρια για το πακέτο για το εμπορικό σήμα που συμπεριλάμβανε και τον κοινωνισμό για το εμπορικό σήμα, τη βασική πράξη που έδινε εκτελεστικέ εξουσίε σε βάση των οποίων υιοθετήθηκε αυτή η αυτό το σχέδιο εκτελεστικές πράξεις. Η Κομισιόν μας ενημέρωσε ότι μελλοντικές συζητήσεις για αυτό το σχέδιο εκτελεστικές πράξεις σε επίπεδο πυρογνωμόνων ε, θα γίνει το Νοέμβριο του 2016. Η Επιτροπή επομένως θα επανέλθει στο θέμα αυτό το Νοέμβριο. Η γραμματεία της Επιτροπής έχει λάβει ο ένα σχέδιο πράξης που βασίζεται στην ίδια βασική πράξη. Οι συντονιστές έχουν επίσης διορίσει την κυρία Βίξτρομ εισηγήτρια για αυτό το σχέδιο ε, της πράξης και τα μέλη θα ενημερωθούν όταν θα έχει γίνει επίσημη παραπομπή στο Κοινοβούλιο. Αυτό για το σημείο 12. Λίγο από σχόλια. Καθώς λοιπόν ο κύριος Τύρα δεν έχει έρθει ακόμη, να περάσουμε στο σημείο 31. Έχει να κάνει με την ερμηνεία και την εφαρμογή της Διοργανικής Συμφωνίας για την καλύτερη νομοθεσία. Εγώ είμαι ο εισηγητής ή ο συνεισηγητής, για να το πω καλύτερα, για τη δική μας Επιτροπή. Στις 3 Οκτωβρίου 2016, η ομάδα εργασία για την ερμηνεία και την εφαρμογή της ε, Διοργανικής Συμφωνίας για την καλύτερη νομοθεσία, συνεδρίαση για τέταρτη φορά, η ομάδα εργασία επικεντρώθηκε στα κριτήρια καθορισμού μεταξύ των κατοξιδότηση και των εκτελεστικών πράξεων και είχε μια ανταλλαγή απόψεων με τους δύο διαπραγματευτές για το Κοινοβούλιο, τους κυρίους Σάιερ και Κορμπέτ. Τόνισα ότι το κεφάλαιο 5 της νέας διοργανικής συμφωνίας ήταν και επιτυχία αλλά και μια χαμένη ευκαιρία. Είναι σημαντική επιτυχία ότι οι εμπειρογνώμονε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα εμπλέκονται στην προετοιμασία των κατοξιδότηση πράξεων ε, ισότιμα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών. Παρ' όλα αυτά, το γεγονός ότι η Κομισιόν απαιτείται να διαβουλεύεται με εθνικούς εμπειρογνώμονες ε, καταλήγει στο να κάνει παρόμοια την όλη διαδικασία, αν όχι ταυτόσιμη σε αυτή που υπάρχει για την προετοιμασία των εκτελεστικών πράξεων. Αυτό μπορεί λοιπόν να θολώσει τις διαφορές μεταξύ των δύο τύπων πράξεων. Ο κ. Κορμπέτ συμφώνησε ότι σχετικές διατάξεις της Διοργανικής Συμφωνίας συνιστούσαν πρόοδο όμως και παραχωρήσεις που θα μπορούσαν να θολώσουν την διάκριση μεταξύ κατεξουσιοδότης και εκτελεστικών πράξεων. Παρ' όλα αυτά, το σημερινό κείμενο θα πρέπει να ενθαρρύνει το Συμβούλιο να δεχτεί τη συμπερίληψη των κατεξουσιοδότης πράξεων πιο συχνά. Ο κ. Σαΐρ υπενθύμησε τη σημασία της ευθυγράμμισης μεταξύ των δύο ειδών πράξεων και της, συγγνώμη, του καθορισμού ορίων μεταξύ των δύο πράξεων και της ευθυγράμμισης με τις διατάξεις επιτροπολογίας. Οι διαπραγματεύσεις για τα κριτήρια του καθορισμού θα έπρεπε να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν βάσει της έκθεσης της 25ης Φεβρουαρίου 2014. Ο κύριος Σάιερ αναγνώρισε ότι προκειμένου να ξεπεραστεί μια στάσιμη κατάσταση δέχτηκε το Κοινοβούλιο υποχρεωτική διαβούλευση με του εμπειρογνώμονε στην προετοιμασία των κατεξουσιοδότηση πράξεων. Αυτό τώρα θα πρέπει να οδηγήσει το Συμβούλιο να δεκτεί πιο εύκολα τι κατεξουσιοδότηση πράξει. Αυτά από μένα. Θα ήθελε κάποιος το λόγο. Όχι, ο κύριος Αίρε Επομένως, ολοκληρώνεται και αυτό το σημείο. Uh, λοιπόν, καθώς ο κύριος ε, Ντυρά δεν έχει εμφανιστεί ακόμη, θα πρότεινα να κάνουμε ένα διάλειμμα μέχρι τις 4 και 4 έτσι ώστε να μπορέσει να έρθει ο κ. και να πάρει το λόγο και κατόπιν θα συνεχίσουμε με τη συνεδρίαση και κλεισμένων των θηρών έτσι όπως ε, βλέπετε στην ίδια διάταξη. Τα λέμε στις 4 και 4.